καλωσορίσω όλους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Mam nadzieję, że odpoczęliśmy, chociaż te wakacje były inne. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε όλοι στις ε, διακοπές. Και Σίγουρα άλλαξαν πολλά πράγματα σε σχέση με το παρελθόν ε, για τις ε, διακοπές μας. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και με στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Ήμουν σε διαρκή επαφή με την Πολωνική Προεδρία, του εκπροσώπους της Πολωνικής Προεδρίας, λόγω της κρίσης, ε, που είναι ένα θέμα φυσικά το οποίο απασχολεί όλους μας, ε, στις 29 Αυγούστου, όπως ξέρετε, ε, διοργανώσαμε μια ειδική επιτροπή της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με τον κύριο Όλι Ρένε, τον κύριο Τρισέ, τον κύριο Γιούγκερ, και τον Υπουργό Ροστόφσκι. Ο κύριος Μπαρόζο σύντομα θα καταθέσει προτάσεις και ο Πρωθυπουργό Γιούνκερ, πρόεδρος της, του Eurogroup, ε, θα ε, κάνει τις εισηγήσεις του επίσης κατά το μήνα Σεπτέμβρη. Το καλοκαίρι ε, σταμάτησαν οι εχθροπραξίες ε, στην ε, Λιβύη και με ικανοποίηση μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ταχθεί στο σωστό, συνταχθεί στο σωστό στρατόπεδο από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τα ψηφίσματά μας και τώρα αυτό που απομένει είναι να βοηθήσουμε το λαό της Λιβύης να ανοικοδομήσει τη χώρα του, να το συνοδεύσουμε σε, αυτήν, σε αυτό το δρόμο προ τη δημοκρατία έχει προβλεφθεί συζήτηση για αυτό το θέμα και άρα θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας. Ο κύριος Φερχόφστατ μου ζητάει το λόγο. Παρακαλώ, ένα διαδικαστικό, Πρόεδρε, διότι αναφερθήκατε στην κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Ποια πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβουμε, αληθεύει, ότι θα σανθείτε αύριο με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον κύριο Μπερλουσκόνη, εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, η σύσκεψή σας θα φέρει επιπίου θέματος. Ε, δεν ξέρω, δεν θέλω να συζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους συγκαλέσατε τη σύσκεψη. Ε, ε, ρωτώ μόνο αν αληθεύει και αν αληθεύει ότι θα τον συναντήσετε, δεν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να του ζητήσετε να πάει και στην αρμόδια για αυτό το πρόγραμμα λιτότητας επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ο κύριος Παπανδρέου αυτό έκανε. Ήρθε στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει το πρόγραμμα λιτότητας ε, και απευθείας, απευθείας πήγε στην Επιτροπή Κρίζ για να εξηγήσει το σχέδιό του και ήταν πάρα πολύ επικοδομητική συνεδρίαση. Οπότε ρωτώ, δεν ξέρω για ποιους λόγους έγινε αυτό, για ποιους λόγους έρχεται ο κύριος Μπερλουσκόνη αύριο, αλλά αν έρχεται Γι' αυτό το πρόγραμμα λιτότητα ε, ζητώ επίσημα να παραστεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για να μα παραθέσει το πρόγραμμά του. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρεμπέκα ε, Θα ήθελα να πω ότι στηρίζω την παρέμβαση του συναδέλφου κ. Φέρχοφστατ εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα. Αλλά θέλω να θέσω το ερώτημα κατά πόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τελικά κάνουν μια χάρη στον Μπερλουσκόνη να τον δουν μια μέρα όπου ε, όπου θα πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο λόγω της δίκης εναντίον του για εκπόρνευση ανηλίκου. Κυρίες και κύριοι, αν ε, δίνουμε μια αξία στο να ληφθούν οι θεσμοί στην Ιταλία σοβαρά και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, δεν θα έπρεπε εμείς να επιλέξουμε μια διαδικασία ε, με το Μπερλουσκόνη που να μην του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ε, θα ήθελα να παρακαλώ τον κύριο Μπούζε και τον κύριο Παρόζο να σκεφτούν κατά πόσο μια τέτοια ημερομηνία όπου εκρεμεί μια δίκη κατά του κυρίου Μπερλουσκόνη στην Ιταλία θα πρέπει να συναντηθούμε, ε, είναι δεδειγμένα να συναντηθούμε μαζί του και να γίνουν αυτές οι συζητήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάρμς, ο κύριος Μάουρο signor ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. σημειώνω την πρόταση του κυρίου Φερχόφστατ που είναι απόλυτα λογική κατά την άποψή μου. Είμαι βέβαιος ότι αν το κοινοβούλιο προσκαλούσε τον ε, Ιταλό Πρωθυπουργό από οποιασδήποτε συνθήκες είμαι βέβαιος, παραλαμβάνω, ότι όπως δείχνει και η αυριανή επίσκεψη του κυρίου ε, Μπερλουσκόνη, η Ιταλική κυβέρνηση θα έκανε ό,τι μπορούσε για να ε, γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά αυτό που λέει η κυρία Χάνς με εκπλήσει. Τώρα, τον κύριο Μπερλουσκόνη μπορεί κανείς να τον συμπαθεί ή όχι. Εξακολουθεί να είναι όμως ο Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Ο Πρωθυπουργό μιας χώρας που ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή η χώρα αυτή. Η ομάδα των ε, Πρασίνων δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να ε, εγκαλεί τον κύριο Μπερλουσκόνη ή οποιονδήποτε άλλον και να δίνει μαθήματα δημοκρατίας. Και υπό το πρίσμα της επίσκεψης του κυρίου Μπερλουσκόνη ε, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να ζητήσουμε να συναντηθεί και με τους επικεφαλείς των ομάδων. Κύριε Πρόεδρε, ίσως ε, να έρθει ο κύριος Μπερλουσκόνη αύριο. Δεν ξέρω, αυτό μου είπε ο συνάδελφος κύριος Μάουρο. Γιατί θέλει να είναι ο πρώτος ο οποίος θα συγχαρεί τον κύριο Σούλτς στον αυριανό του διορισμό. Θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, κύριε Πρόεδρε, το δικό μου ενδιαφέρον είναι διαφορετικό. Α, την Τετάρτη στις 2-3.30 ε, λαμβάνει χώρα μια ανοιχτή για όλους συνεδρίαση της συνδιάσκεψης των Προέδρων εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας. Θα πρέπει να συντομεύσουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ε, για να λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση. Μέχρι τώρα η αίθουσα της Ολομέλειας ε, προορίζονταν μόνο για επικεφαλής κυβερνήσεων και νομίζω ότι είναι τρομερό να πρέπει να συντομεύσουμε τη δική μας συνεδρίαση γιατί κάποιος θέλει να κάνει μια ακρόαση ενός υπαλλήλου σε αυτή την αίθουσα. Πρώτη φορά συμβαίνει ακρόαση υπαλλήλου σε αυτή την αίθουσα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να γίνει συζήτηση για την κρίση του χρέους ολόκληρο το απόγευμα όπως έχει προβλεφθεί. Αυτό είναι ζήτημα της διάσκεψης των Προέδρων λέει πρόεδρο, Σας ευχαριστώ πάντως ε, που μας επιστήσατε την προσοχή σε σχέση με το πρώτο θέμα το οποίο αναφέρατε. Κυρίες και κύριοι, εξ όσων γνωρίζω και με βάση τις πληροφορίες που έχω, ο Πρωθυπουργό κύριος Μπερλουσκόνη δεν ε, έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης Δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, ήθελα να περάσω στην επόμενη ανακοίνωσή μου. Αύριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ξέρουμε ότι θα αναφέρουμε αύριο τον πρόεδρο της Πολωνίας. Ξέρουμε ότι η Πολωνία ασκεί την προεδρία. Ο πρόεδρος Χακομορόσκι θα, θα έρθει εδώ και θα έχουμε μια πανηγυρική συνεδρίαση το μεσημέρι. 15 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα της δημοκρατίας. Τη δημοκρατία πρέπει να την προστατεύουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό πράττει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι και το πλέον δημοκρατικό από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα σας δώσω τώρα τι επόμενε πληροφορίε στα αγγλικά. Θέλω να καταδικάσω επισήμως ε, τις βιαιότητες ε, της ε, Δευτέρας Ιουλίου ε, κατά του συναδέλφου μας Ευρωβουλευτή Αγιάτα Καρίμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ιδιωτική του κατοικία έπεσε θύμα επίθεση, 15 μελών μιας εξτρεμιστική οργάνωσης μπήκαν ε, στην ε, ε, κατοικία του φέροντας αντισλαμικά πανό τον έβριζαν και μάλιστα φωτογράφησαν, μαγνητοσκόπησαν και το σπίτι του και ήταν μέσα και η οικογένειά του εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο πάντοτε και πάντοτε πρέπει να καταδικάζουμε περίφραστα τέτοια συμβάντα, ιδίως όταν ε, πρόκειται για ε, εγκλήματα μίσους, ε, τα οποία πλήττουν την ελευθερία έκφρασης ευρωβουλευτών. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Καρίμ έχει λάβει εντολή σε δημοκρατικές εκλογές από τους Βρετανούς πολίτες. Οποιαδήποτε δηλαδή, λοιπόν επίθεση κατά του προσώπου του ή της οικογένειάς του είναι και πλήγμα κατά της δημοκρατίας και των ε, εκλογέων του. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο κύριος Καρίμα να προστατευτεί, να μπορεί να ασκήσει τις ελευθερίες του, την ελευθερία έκφραση, την ελευθερία λόγου, χωρίς να δέχεται απειλές και να μπορέσει να επιτελέσει το πολιτικό του έργο ως ε, δημοκρατικός ε, εκλεγμένος πολιτικός. Εξού λοιπόν καλό να στηρίξουμε τον ε, κύριο Καρίμ. Έχω γράψει μια επιστολή προς τον κύριο Κάμερον και θέλω δημοσία σήμερα να επαναλάβω ε, κύριε Καρίμ σε εσά προσωπικά την απόλυτη υποστήριξή μου καθώς και σε όλους όσους πέφτουν θύματα διακρίσεων. Το Κοινοβούλιο είναι πάντοτε στο πλευρό σας. Προασπίζουμε πάντοτε τις κοινέ μας αξίες ως Κοινοβούλιο. Συναντήθηκα προσωπικά πριν από δύο τρεις εβδομάδες με τον ε, κύριο Κάριμ, πεντής διακοπές. Ε, is another point of order; υπάρχει διαδικαστικό, κύριοι Λινάτη, παρακαλώ. Sul punto precedente, la visita del presidente Berlusconi a questa istituzione προηγούμενο σημείο για την επίσκεψη του Πρόεδρου Μπερλουσκόνη στο Κοινοβούλιο. Ε, καταλάβαμε όλοι ότι έχουν υποθεί διάφορα υπερβολικά πράγματα για αυτή την επίσκεψη. Μετά τη δική σας διευκρίνηση καταλαβαίνουμε ότι δεν προβλέπεται επίσημη επίσκεψη του Προέδρου ε, στο Κοινοβούλιο. Ωραία. Εάν θα τον συναντήσετε λοιπόν, ποιο θα είναι το καθεστώς αυτής της συνάντησης. Η κοινή γνώμη στην Ιταλία θεωρεί ότι πρόκειται για ε, φαρσοκομωδία, διότι αύριο έπρεπε να παραστεί ενώπιον της εισαγγελία ο κύριος Μπερλουσκόνη. Μάριο Μάουρο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, θα μπορούσατε κάλλιστα να μας ενημερώσετε ενδελεχέστερα για τους όρους που διέπουν αυτή τη συνάντηση και έτσι θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την φάρσα διότι ε, δέχεται επιθέσεις η Ιταλική κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν έχει ε, καμία σχέση με το αντικείμενο της επίσκεψης του κ. Μπελουσκόνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι δικαστέ στην Ιταλία είπαν ότι θα ορίσουν άλλη ημερομηνία. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Πρόεδρος, ε, εξήγησα και προηγουμένως περί τίνος πρόκειται. Δεν έχει υποβληθεί αίτημα για επίσημη επίσκεψη από πλευράς του κ. Μπερλουσκόνη. Ενδέχεται να έρθει αύριο στο Κοινοβούλιο. Ενδέχεται. Δεν μπορώ να αποκλείσω μία επίσκεψη απλή, για λόγους ευγενείς, για λόγους τυπικούς, αλλά επίσημη επίσκεψη δεν πρόκειται να γίνει. Ενδέχεται αύριο δεν να έρθει και ο πρόεδρος ε, της ε, Πολωνίας. Αύριο θα είμαι ιδιαίτερα απασχολημένος ως εκ τούτου γιατί θα πρέπει να υποδεχθώ τους προσκεκλημένους μας δεν ε, δίναμε να προσθέσω στο πρόγραμμά μου άλλη επίσκεψη, όπως παραδείγματος χάρη μία επίσκεψη του κυρίου Μπερλουσκόνη. Έτσι έχει η κατάσταση. Θα μπορούσαμε, συνάδελφοι, να ε, σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί σας είπα όλα αυτά που ξέρω. Ποιος άλλος θέλει το λόγο, ένα λεπτάκι. Κανείς, λαμπρά. Μπορούμε να ε, σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση και να προχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι, έχω διάφορες ανακοινώσεις. Μετά την τελευταία σύνοδό μας ε, που έληξε στις 7 Ιουλίου, ε, στις 7 Ιουλίου ε, εγκρίθηκαν και τα πρακτικά, δεν έχετε σχόλια βλέπω.